Ladies and gentlemen, dear colleagues. Συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε. Περνάμε στο σημείο 9 της σήμερης διάταξης της ε, Επιτροπής ε, Εξωτερικών Υποθέσεων. Σε συνεργασία με την Επιτροπή Ανάπτυξης έχουμε εδώ τον πρόεδρο Τόμας Τομπέ στο βήμα. Καταρχάς, ε, συνάδελφοι, να καλωσορίσουμε τον ε, κύριο Ταγκέζε Τσάβο, πρόεδρο του Κοινοβουλίου της Αιθιοπίας και ε, να καλωσορίσουμε και τον πρέσβη Άμπαε και τον κύριο Τέσφεϊ Ντάμπα, σωστά το, σωστά, ε, σωστά το είπα το όνομα, που είναι πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Αιθιοπικού Κοινοβουλίου. Σας καλωσορίζουμε όλους. So, um, the only Ethiopian word I know is Τένα Γίστελιν. Τένα Είναι η μόνη λέξη στα αιθιοπικά που ξέρω. Ε, καλωσορίσατε νομίζω ότι σημαίνει. Σωστά τα λέω. Λοιπόν, ποιο θα μπορούσε να φανταστεί όταν σχεδιάζαμε αυτή τη συνάντηση ότι θα ερχόταν σε τόσο κατάλληλη στιγμή. Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς να σας ε, εκφράσουμε τα θερμότατα συγχαρητήριά μας για την ε, απονομή ε, στον κύριο Πρωθυπουργό τον Άβη Άμετ του Νόμπελ Ειρήνης για τις προσπάθειες που κατέβαλε για τη διεθνή συνεργασία και τη διεθνή ειρήνη. Συνέβαλε σημαντικότατα στην επίλυση του ζητήματος ε, με τα σύνορα με την ε, ε, γειτονική Ερυθρέα, που είναι και ένα ζήτημα που μας έχει απασχολήσει. Θέλουμε λοιπόν να διαβιβάσετε τα συγχαρητήριά μας στον Πρωθυπουργό σας Είναι λοιπόν πολύ κατάλληλη στιγμή, γιατί και οι δύο επιτροπέ μα με την Επιτροπή ανάπτυξη είναι κοινή συζήτηση αυτή που θα γίνει, ε, σχεδιάζουμε να κάνουμε σύντομα μια επίσκεψη στη χώρα σα και θέλουμε Τώρα να ακούσουμε από εσά ε, ποια είναι η αξιολόγησή σα, ποια είναι η εκτίμησή σα για την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην Αιθιοπία και για το μέλλον τη ε, χώρα αλλά και τη ευρύτερη περιοχή. Θα δώσω το λόγο στον συνάδελφο, τον κύριο Πέτρε Ταμπού, και στη συνέχεια θα, το μπε και στη συνέχεια θα ε, προχωρήσουμε στην ε, συζήτηση. Ευχαριστώ κύριε Μακάλιστερ, σας ε, καλωσορίζω και εκ μέρους της Επιτροπής Ανάπτυξης, κύριε Πρόεδρε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Από την σκοπιά της δικής μου Επιτροπής, της Επιτροπής Ανάπτυξης, η, η είναι ένας εξαιρετικός εταίρος λόγω της, του μεγέθους της, της των ε, μεγάλων προκλήσεων που αντιμετωπίζει όσον αφορά την ανάπτυξη, αλλά και λόγω της ε, κλίμακας ε, της ευρωπαϊκής συνεργασίας μαζί σας, της αναπτυξιακής συνεργασίας, λόγω και της ιδιαίτερης οικονομικής ανάπτυξης που έχετε επιτύχει τα τελευταία χρόνια και λόγω της ραγδαίας προόδου που έχετε σημειώσει στον τομέα της οικονομικής ανάπτυξης. Θέλω να αναφέρω και τις τολμηρές ε, και καινοτόμες ε, νέες πολιτικές που εισήγαγε ο κύριος Σαμπάιτο τους τελευταίους 18 μήνες που την χάνουν ε, της ελπίδας αλλά και του θαυμασμού όλων μας. Ωστόσο, όταν σε μια τέτοια χώρα με τόση ποικιλομορφία ανοίγει η δημοκρατική διαδικασία είναι πολύ σημαντικό να προστατευτεί και η συνοχή και να προστατευτούν και οι δημοκρατικές πρακτικές και διαδικασίες. Είναι λοιπόν ελπίδα και αγωνία μαζί αυτή που χαρακτηρίζει εμάς ε, παρακολουθώντας τις χώρες σας. Θέλουμε να σας ευχηθούμε κάθε επιτυχία στη μετάβαση αυτή και θέλω να σας πω ότι σε μόλις δύο εβδομάδες θα έχω την ε, τιμή να είμαι επικεφαλής αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της Επιτροπής Ανάπτυξης προς την, ε, στην Αιθιοπία, στη χώρα σας. Πριν από εμά, λέει ο κύριος Μακάλιστερ, βεβαίως. Εμείς ε, είχαμε προβλέψει σωστά τα πράγματα, ξέραμε τι θα επερχόταν και θέλουμε αυτή η επίσκεψή μας να συμβάλλει σε μεγαλύτερη κατανόηση των δύο πλευρών και πραγματικά εκφράζω την ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίησή μου που θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε αυτό το διάλογο μαζί σας και πλέον προσβλέπουμε βεβαίως και στον, ε, στην ομιλία στα όσα έχει να μας πει ο κύριος Πρόεδρος. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ για τα θερμά σας λόγια. Ε, πρόεδρε της Επιτροπής Ανάπτυξη και της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, αξιότιμα μέλη των Επιτροπών, αξιότιμοι ευρωβουλευτές. Η αντιπροσωπεία μου θα ήθελε να ευχαριστήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την υποδοχή εδώ σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά και για τη θερμότατη ε, ε, υποδοχή που μας επιφυλάξατε. Είναι πραγματικά μεγάλη τιμή για την αντιπροσωπεία μου να βρισκόμαστε σήμερα εδώ μαζί σας για να συζητήσουμε τα πολύπλευρα ε, ζητήματα και τις εξελίξεις και τις μεταρρυθμίσεις που βρίσκονται σε εφαρμογή αυτή τη στιγμή στην Αιθιοπία και στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και ε, προκειμένου να γίνει μια ανταλλαγή απόψεων για διμερή και περιφερειακά ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος. Όπως γνωρίζετε ίσως, από, τον, από την εκλογή του κυρίου Αμπιάματ ως Προέδρου του κυβερνώντος κόμματος του IPRDF και το 2017 η Αιθιοπία έχει ξεκινήσει μια μαζική ε, διαδικασία μεταρρύθμισης, μετασχηματισμού πολιτικού, ε, ε, στον πολιτικό, τον οικονομικό και το δικαστικό τομέα. Πολιτικά η κυβέρνηση έχει λάβει θεμελιώδη μέτρα για να εξασφαλιστεί το άνοιγμα του πολιτικού χώρου με τρόπο που θα εξασφαλίζει ίσους όρους ε, για όλα τα πολιτικά κόμματα και τους πολιτικούς φορείς. Και στο πλαίσιο αυτό, χιλιάδες πολιτικοί κρατούμενοι, δημοσιογράφοι ε, έχουν ε, λάβει χάρη και έχουν απελευθερωθεί από τις φιλιακείς. Ε, ομάδες εξορίστων των πολιτικών έχουν ε, προσκληθεί να επιστρέψουν στη χώρα για να συμβάλλουν με ειρηνικό τρόπο στην, στον μετασχηματισμό της χώρας. Και τρεις ε, ένοπλες ομάδες που θεωρούνταν ε, τρομοκρατικές ε, ομάδες αφαιρέθηκαν από τον κατάλογο πλέον. Θέλουμε αυτές οι μεταρρυθμίσεις να κατοχυρωθούν και συνταγματικά. Έχουν γίνει πολλές νομικές μεταρρυθμίσεις, δημιουργήθηκε γραφείο Γενικής Εισαγγελίας και υπάρχει πλέον και μια ομάδα 13 νομικών εμπειρογνωμόνων που εξετάζουν ε, τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος και πρόκειται να αναπτύξουν συστάσεις για ολοκληρωμένες ε, αναθεωρήσεις συμπεριλαμβανομένων και τροποποιήσεων νόμων αλλά και την θέσπιση νέων νόμων. Επίσης, αναθεωρείται ο νόμος για την κοινωνία των πολιτών, για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ο εκλογικός νόμος, που έχουν, ο οποίος πλέον έχει αναθεωρηθεί και επικυρωθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ο νόμος ε, κατά της ε, τρομοκρατίας επίσης είναι ένας από τους νόμους που βρίσκονται υπό αναθεώρηση. Η κυβέρνηση της Αιθιοπίας επίσης έχει λάβει μέτρα για την απελευθέρωση της οικονομίας και την ιδιωτικοποίηση μερική ή ολική κρατικών επιχειρήσεων ε, με, που συνέβαλαν σημαντικά στην, ε, σε μακροοικονομικές ανισορροπίες στη χώρα. Έχουμε λοιπόν μια ε, ατζέντα οικονομικών μεταρρυθμίσεων που αποσκοπεί στο να ε, ε, γίνουμε μια χώρα μεσαίου εισοδήματο έως το 2030 μέσω της ε, οικοδόμησης της ε, δημιουργίας ενός ε, ισχυρού ιδιωτικού τομέα μέσω της κοινοτομίας η οποία μπορεί να μας ε, οδηγήσει στην, στον εξυγχρονισμό και την αύξηση της γεωργικής παραγωγής. Επίσης, η, δημιουργήθηκε Εθνική Επιτροπή υπό τον Πρωθυπουργό που ε, εξασφαλίζει την, ε, ένα φιλικό προς τις επιχειρήσεις περιβάλλον γενικά. Και από αυτή την άποψη οι βασικοί στόχοι του προγράμματος μεταρρυθμίσεων δημιουργούν ευκαιρίες απασχόλησης για τους νέους μας και θέτουν ε, επικεφαλής της διαδικασίας βιομηχάνησης και εξυγχρονισμού των ιδιωτικών τομέα. Επίση, η ενίσχυση των γυναικών ισότητα των δύο φύλων είναι επίση ένα τομέα στον οποίο η κυβέρνηση τη Αιθιοπία έχει εστιάσει την προσοχή τη. Όπω ίσω έχετε γνωρίσει, τα μισά μέλη τη κυβέρνηση ε, τη ε, Αιθιοπία είναι γυναίκε. Καταλαμβάνοντα ε, σημαντικότατε θέσει όπω είναι η Προεδρία, το Ανώτατο Δικαστήριο, η, Επιτροπή, ε, η Εκλογική Επιτροπή επίσης έχουν όλες επικεφαλής γυναίκες και από τις 10 μόνιμες κοινοβουλευτικές επιτροπές, 6 από αυτές έχουν προέδρους γυναίκες στο Κοινοβούλιο της Αιθιοπίας. Αξιότιμα μέλη των Επιτροπών, κύριε και κύριοι, η Αιθιοπία προετοιμάζεται για εθνικές βουλευτικές εκλογές που θα γίνουν το 2020. Και από αυτή την άποψη ε, ε, λαμβάνονται τα αναγκαία θεσμικά και δημοκρατικά μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα γίνουν εκλογές ειρηνικές, δημοκρατικές, νόμιμες. Και για το σκοπό αυτό έχει αναδιοργανωθεί και η Εθνική Εκλογική Επιτροπή πέρσι με τρόπο ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ευθύνες της με ε, τις μέγιστες δυνατές ε, δυνατότητες και τη μέγιστη δυνατή αξιοπιστία. Αναθεωρήθηκε ο εκλογικός νόμος και επικυρώθηκε από το Κοινοβούλιο και οι αναγκαίες συζητήσεις ε, και διαβουλεύσεις έχουν γίνει με όλους τους εμπλεκόμενους και ενδιαφερόμενους φορείς συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων των κοινων... της κοινωνίας των πολιτών, των μέσων μαζικής ενημέρωσης, της κοινής γνώμης και των πολιτικών κομμάτων. Η κυβέρνηση ξεκίνησε έναν ανοιχτό διάλογο με όλα τα πολιτικά κόμματα και υπέγραψε έναν κώδικα δεοντολογίας ο οποίος θα διέπει τις συμπεριφορές και τις δραστηριότητες όλων των πολιτικών κομμάτων στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές του 2020. Αγαπητά μέλη των Επιτροπών, κυρίες και κύριοι, η συνεχιζόμενη αλλαγή στην Αιθιοπία έχει ξεκινήσει και μια ευρύτερη διαδικασία ε, μεταρρυθμίσεων στο κέρας της Αφρικής. έχει ξεκινήσει πραγματικά μια νέα εποχή συνεργασίας στην περιοχή μας. Η Αιθιοπία συνέβαλε στο μέτρο των ευθυνών της στην, ε, στον τερματισμό των βιοπραγιών στο Σουδάν. Επίσης συμμετέχει στην ε, ειρηνευτική διαδικασία στο Νότιο Σουδάν. Έπαιξε σημαντικό ρόλο, επικοδομητικό ρόλο στην ε, βοήθεια προς την Σομαλία για την καταπολέμηση των Νισαβά και θεωρεί ότι ε, είναι σημαντική η, συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ε, διεθνούς κοινότητας στην επίλυση των προβλημάτων της Σομαλίας. Κυρίες και κύριοι, η, η Αιθιοπία περνά μια πραγματική αναγέννηση και στην ηλεκτροπαραγωγή. Μιλάμε για μια χώρα όπου 60% του πληθυσμού δεν έχει πρόσβαση σε, ηλεκτρικό ρεύμα. Δείξαμε την προσήλωσή μας στη δημιουργία ενός πολυμερούς νομικού καθεστώτος όσον αφορά την αξιοποίηση ε, της λεκάνης του, Νείλου, του ποταμού του Νείλου καταβάλαμε μεγάλες προσπάθειες προκειμένου να επιληθούν τεχνικά προβλήματα που αντιμετωπίσαμε. Η Αιθιοπία πιστεύει ακράδαντα ότι μόνο μέσω τεχνικών και επιστημονικών μέτρων μπορεί να επιληθεί το ζήτημα του φράγματος. Είναι απαραίτητο οι τρεις χώρες να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις τους. Αυτό θα κάνει η, η Αιθιοπία όσον αφορά το φράγμα στον ε, ποταμό Νείλο. Κυρίες και κύριοι, η Αιθιοπία βρίσκεται στο μέσο μιας τεράστιας διαδικασίας μετασχηματισμού που, ήτανε, που δεν θα μπορούσαμε να τη φανταστούμε πριν λίγα χρόνια. Έχουμε λοιπόν μεγάλη αισιοδοξία και ελπίδες, αλλά αντιμετωπίζουμε και προκλήσεις, όπως είναι οι σποραδικές συγκρούσεις εδώ και εκεί που έχουν οδηγήσει στον εκτοπισμό χιλιάδων ανθρώπων. Η κυβέρνηση προσπαθεί να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της, και για την επιστροφή των εκτοπισμένων, κάτι που έχει ήδη σε μεγάλο βαθμό επιτευχθεί, αλλά και για να καταπολεμηθούν τα γενεσιουργά αίτια αυτών των προβλημάτων. Οι εποχές ε, αλλαγών και μετασχηματισμών ε, συνοδεύονται πάντοτε και από συνειδητοποίηση του μεγέθους ε, των προβλημάτων και των προκλήσεων που αντιμετωπίζει κανείς. Εμείς όμως είμαστε αισιόδοξοι ότι θα ξεπεράσουμε όλα τα εμπόδια που αντιμετωπίζουμε και ε, σας καλώ να μας υποστηρίξετε και να επιδείξετε κατανόηση ως εταίροι μας εδώ στην Ευρώπη. Τέλος, Όσον αφορά τι ε, σχέσει ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αιθιοπία, θα θέλαμε για άλλη μια φορά να ε, εκφράσουμε την προσήλωσή μας και την επιθυμία μας να έχουμε μια επικοδομητική συνεργασία, μια αγώνιμη συνεργασία προς όφελος των αμοιβαίων μας συμφερόντων. Σας ευχαριστώ για το χρόνο και για την προσοχή σας. Thank Σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε ε, ένα μισάωρο περίπου για ανταλλαγή απόψεων και θα ήθελα να δώσω το λόγο στους πρώτους συναδέλφους που ζήτησαν. Παρακαλώ να περιοριστείτε στα τέσσερα λεπτά. Ξεκινάμε το Μιχαήλ Γκάλερ από το ΕΛΚ. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ορίσατε και από δική μου πλευρά παρακαλώ να διαβιβάσετε τα συγχαρητήριά μας για το βραβείο Ειρήνης Νόμπελ στον Πρωθυπουργό σας. Βρίσκομαι εδώ και 20 χρόνια στο Κοινοβούλιο και πάντοτε στην, ε, στην ε, Ισομερή Κοινοβουλευτική Συνέλευση που συχνά έχω επισκεφθεί τη χώρα σας το 2004 ε, θυμάμαι ότι μείναμε εκεί για να, ως παρατηρητές ε, το 2005 για τις εκλογές και το 2010 αλλά και το 2015 δεν ήρθαμε γιατί θεωρήσαμε πως δεν άξιζε. Ε, γνωρίζω ότι εντωμεταξύ οι συνάδελφη, ε, η συνάδελφος Άννα Γκόμες που η κυβέρνηση το, η τότε δεν τη συμπαθούσε καθόλου. Εν τω μεταξύ έχει γίνει πολύ ε, καλά δεχτή από τη δική σας κυβέρνηση και ίσως να είναι αυτό σημάδι ενός διαφορετικού πολιτικού κλίματος. Έχω όμως ε, δύο διαφορετικές ερωτήσεις. Η διαδικασία στην οποία αναφερθήκατε και αναφερθήκατε μάλιστα και στις επόμενες εκλογές του 2020, αυτές οι Αλλαγέ είναι για όλους, δηλαδή συμπεριλαμβάνονται και τα κόμματα της αντεπολίτευση, η κοινωνία των πολιτών και όλοι όσοι θα ήθελαν να γίνουν καλύτερες εκλογές την επόμενη φορά και όχι μόνο εκλογές όπου το ίδιο κόμμα θα κερδίσει πάλι. Μπορείτε λίγο να μας εξηγήσετε. Γιατί θυμάμαι ότι τέτοιες συζητήσεις είχαμε ήδη πριν από 10 χρόνια όσον αφορά την εκλογική διαδικασία. Και επίσης ε, παλαιότερα είχαμε και ένα άλλο θέμα, την αρπαγή γης. Την πολιτική δηλαδή όπου καλείς ε, εγκεκριμένους ε, αλλοδαπούς ε, να αρπάξουν τεράστια κομμάτια γης ε, που υποτίθεται ότι ήταν στέρφα και καλλιέργητα, αλλά έχουμε μαρτυρίες από κόσμο που λέει ότι όχι, τα δούλευαν αυτέ τις δούλευαν αυτές τις γης. Τώρα, τι έχετε κάνει για αυτό το ζήτημα και ποιες λεπτομέρειες μπορείτε να μας δώσετε. Ευχαριστώ. Θέλετε να απαντήσετε κάθε ερώτηση χωριστά. Ή να ακούσουμε πρώτα τις ερωτήσεις. Όχι, να προσθέσετε. Ο κύριος Ριβιέρ είναι τώρα από... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να... Διακόπτει ο μιλητής. Merci, Monsieur le Président. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλώς ορίσατε. Και εγώ θέλω εξ ονόματός μου και εξ ονόματος της ομάδας μου να συγχαρώ τον Πρωθυπουργό σας για το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Θα ήθελα να σας ρωτήσω στη διάρκεια αυτών, αυτής της ανταλλαγής απόψεων δύο συγκεκριμένα πράγματα. Το πρώτο είναι ότι η Αιθιοπία υποδέχεται διάφορες ευρωπαϊκές επενδύσεις, ιδιαίτερα όσον αφορά οδικά έργα, κυκλοφοριακό, υποδομές τέτοιου τύπου, αλλά και υπέρ των βελτιώσεων που αφορούν την κοινωνία των πολιτών και την ενίσχυση της δημοκρατικής διακυβέρνησης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάποιες φορές έχει μια εικόνα ε, του ε, σωτήρα, ε, με βάση τα όσα ξέρουμε εμείς εδώ στις δικές μας δυτικές ε, ε, ε, ε, ιδέες. Ε, ε, σας ρωτώ αν όντως όλα αυτά γίνονται και βοηθούν στην Αιθιοπία. Είναι η δική μας εικόνα και ιδέα. Τώρα η δεύτερη ερώτηση αφορούν τους τρομοκράτες μπάμπα στα ανατολικά της χώρας σας. Πέρα από την θρεβερή ιδεολογία που είναι ο λόγος για τις δράσεις τους, πιστεύετε πως ξένες χώρες μπορεί να συμβάλλουν στη δράση τους ε, δηλαδή επηρεάζονται από κάποιο άλλο κράτος ε, ή πρόκειται για μια αυτόνομη τρομοκρατική ε, ομάδα. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Φωτίγκα τώρα, εξ του ECR. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε του Κοινοβουλίου της Αιθιοπίας θα σας ζητούσα να διαβιβάσετε τα συγχαρητήριά μας στον Πρωθυπουργό σας για την απονομή του βραβείου Νόμπελ σε ένα τεράστιο επίτευγμα. Γνωρίζουμε πολύ καλά πως έχουν οι εξελίξεις στη χώρα σας, στην Αιθιοπία, και βέβαια και χάρη στην ε, δραστηριότητα του ε, πρέσβη σα, ο οποίο φροντίζει πάντα να υποβάλει πολύ πλήρε πληροφορίε σε εμά του ευρωβουλευτέ, σε σχέση δηλαδή με τι εξελίξεις ε, στην Αιθιοπία. Γνωρίζουμε δηλαδή όλες αυτέ τις προσπάθειε που έχετε καταβάλει όσον αφορά την οικονομική σταθερότητα και γνωρίζουμε επίση και τα όσα έχουν να κάνουν με την ειρηνευτική διαδικασία. Ένα ζήτημα το οποίο μας είναι ιδιαίτερα προσφυλές σε όλους εμάς που συμμετέχουμε στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ή που συμμετέχουμε στην Υποεπιτροπή Άμυνας και Ασφάλειας. Θα ήθελα πιο συγκεκριμένα να θέσω ένα ερώτημα σε σχέση με την τρομοκρατία και την εξάλληψη της τρομοκρατίας στο κέρας της Αφρικής και πώς συμβάλλει σε αυτό η Αιθιοπία ποια είναι η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα τα οποία έχετε εσείς εντοπίσει. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, θα μπορούσατε να μας δώσετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σε σχέση με τις εξελίξεις που έχετε στις προσπάθειές να μεταρρυθμίσετε το δικαστικό τομέα στη χώρα σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Φωτίγκα. Και έχουμε ακόμα δύο μιλητές, αν συμφωνείτε κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Γκενγκιάση μη εγγεγραμμένος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε του Κοινοβουλίου της Αιθιοπίας, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ σήμερα μαζί μας. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τον Πρωθυπουργό σας γιατί κατάφερε όντως να επιλύσει τη διένεξη αυτή με την Ερυθρέα που είχε κρατήσει 10 ολόκληρα χρόνια. Σημαντικότατο το επίτευγμα αυτό. Το ερώτημά μου όμως έχει να κάνει περισσότερο με ένα άλλο ζήτημα το οποίο μας ανησυχεί όλος ιδιαίτερος και έχει να κάνει με το περιβάλλον. Πρόσφατα στον Διεθνή Τύπο διαβάσαμε άρθρα όσον αφορά την κλιματική αλλαγή και το όλο αυτό ζήτημα που έχει να κάνει με την προσφορά, με την παροχή του ύδατος στη δική σας την χώρα και στην γενικότερη περιφέρεια. Και ξέρουμε ότι η χώρα σε η Αιθιοπία δεν έχει την απαραίτητη υποδομή. Θέλετε να φτιάξετε και αυτό το φράγμα το Renaissance Dam, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό προκειμένου να μπορέσετε να παράσχετε ηλεκτρικό ρεύμα σε ένα μεγάλο μέρος της χώρας σας. Ξέρω όμως ότι προκύπτουν και ζητήματα με, με το Σουδάν και την Αίγυπτο όσον αφορά την παροχή υδατός. Και όσον αφορά τους Αιγύπτους εμπειρογνώμονες, αυτοί λένε ότι 90% του ύδατος έρχεται από τον Νείλο και από την περιοχή που έχει να κάνει με την Αιθιοπία. Και δυστυχώς το διεθνές δίκαιο δεν μας καθοδηγεί επαρκώ για το πώ θα μπορούσαμε να επιλύσουμε τα προβλήματα τα οποία έχουν προκύψει. Ξέρω ότι υπάρχει μια διεθνή συμφωνία όσον αφορά την κατανομή των υδάτων, μια συμφωνία που υπάρχει μεταξύ Αιγύπτου και Σουδάν. Από όσο γνωρίζω όμω δεν έχετε εσεί μια τέτοια συμφωνία με την Αίγυπτο. Θα συμφωνούσατε ότι μια τέτοια συμφωνία θα μπορούσε να αποτελέσει μια λύση για την επίλυση τη σύγκρουση αυτή που σύμφωνα τουλάχιστον με την Αίγυπτο η κρίση αυτή απειλεί με λειψιδρία ή ακόμα και με ξηρασία ένα μεγάλο τμήμα ε, του αγροτικού πληθυσμού τη Αιγύπτου και ενδεχομένω να μην έχουμε και την κατάλληλη παροχή τροφίμων στην περίπτωση αυτή. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αποφύγουμε μία ακόμα σύγκρουση και διένεξη για του λόγου αυτού στην όλη ευρύτερη περιοχή. Πώ πιστεύετε εσεί, κύριε Πρόεδρε ότι θα μπορούσε να επιληθεί το σημαντικότατο αυτό πρόβλημα. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε. Τελευταίος ομιλητή, ο κύριο Χόβενη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε αξιότιμε κύριε Τσάφο, πρόεδρε του Κοινοβουλίου της Αιθιοπίας, αξιότιμοι συνάδελφοι, τα τελευταία χρόνια εξελίξει στην Αιθιοπία καταδεικνύουν ότι το ζήτημα της ασφάλειας είναι πάρα πολύ σημαντικό όσον αφορά την πολιτική ε, αναπτυξιακή συνεργασία στην οποία ακολουθούμε και ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου της Αιθιοπίας μας μίλησε για την κατάσταση της ασφάλειας στη χώρα και πώς η βελτίωση στον τομέα της ασφάλειας έχει οδηγήσει σε μια βελτίωση του οικονομικού επίπεδου της χώρας. Η επίλυση επίσης της διένεξης με την Ερυθρέα αποτελεί ένα πολύ σημαντικότατο επίτευγμα που σαφώς έπρεπε να βραβευθεί με το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Και ξέρετε πολύ καλύτερα εσείς από ότι εμείς ότι ακόμα απομένουν πολλά τα οποία πρέπει να γίνουν. Θα ήθελα πάντως και εγώ με τη σειρά μου να συγχαρώ τον Πρωθυπουργό σας, Άμπι Αχμέτ, για τη βράβευση αυτή. Αν λάβουμε τώρα υπόψη μας την κατάσταση σε χώρες γύρω από την Αιθιοπία, όπως το Σουδάν, το Νότιο Σουδάν και η Σομαλία, εκεί συνειδητοποιούμε ότι υπάρχουν νέες μεταναστευτικές ροές που επηρεάζουν την Αιθιοπία. Και βλέπουμε ότι ε, η όλο και βελτιωνόμενη οικονομική κατάσταση Αιθιοπίας την έχει καταστήσει μια χώρα προορισμού για πάρα πολλούς μετανάστες και πρόσφυγες. Ήδη όμως έχετε υποδεχθεί ένα εκατομμύριο πρόσφυγες, αν δεν κάνω λάθος. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι η ακόλουθη. Η κατάσταση όσον αφορά την ασφάλεια των γειτονικών χωρών ενδεχομένως να αποσταθεροποιήσει την Αιθιοπία. Πώς διαχειρίζεστε εσείς την όλη κατάσταση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Πρόεδρε του Κοινοβουλίου της Αιθιοπίας, ακούσατε τις ερωτήσεις από τους συναδέλφους. Θα σας δώσω τώρα το λόγο, αλλά πρέπει να σας ενημερώσω ότι θα πρέπει να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση στις 5.30, σε 20 λεπτά δηλαδή. Ευχαριστώ πολύ για τις πολύ ενδιαφέρουσες αυτές επικοδομητικές σας ερωτήσεις. και θα ήθελα ειλικρινά να σε ευχαριστήσω για όλα αυτά τα θερμά λόγια που είπατε για τον Άμπι Αχμέτ των τον ε, Πρωθυπουργό μας και όταν επιστρέψω στην Αιθιοπία θα του διαβιβάσω τα θετικά σε αυτά λόγια τα οποία προέρχονται από την Επιτροπή ε, Εξωτερικών Υποθέσεων. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ για τα θερμά σας λόγια. Όσον αφορά τώρα τις ερωτήσεις, η πρώτη από τον πολύ στενό μου φίλο, τον κύριο Γκάλερ, τον οποίο τον γνωρίζω πάρα πολύ καλά από τη συνεδριά της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης. Για πάρα πολλά χρόνια γνωριζόμαστε και συνεργαζόμαστε και όπως σας είπα όλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη διαδικασία της ένταξης, της ενσωμάτωσης, στον πολιτικό τομέα δηλαδή, μια πολιτική ολοκλήρωση χωρίς αποκλεισμούς, αυτό το ανέφερα και στην εισαγωγική μου παρέμβαση. Πολλέ είναι οι δράσει τη κυβέρνηση, για παράδειγμα η απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων. Και έχουμε και μια ισότιμη εκπροσώπηση όλων των πολιτικών κομμάτων. Ακόμα και για τα πολιτικά εκείνα κόμματα τα οποία επιβαρύνονταν από κάποιες κατηγορίες τρομοκρατικών επιθέσεων το ότι δημιουργήσαμε ένα θετικό επικοδομητικό πνεύμα συνεργασία, αυτό είχε πολύ θετικές συνέπειες. Όταν ε, συστήσαμε το εκλογικό συμβούλιο, συμμετείχαν όλα τα πολιτικά κόμματα από όλο το πολιτικό φάσμα της χώρας. Όπως σας είπα, είναι πέντε τα μέλη και η επικεφαλής του Συμβουλίου αυτού ήταν στο εξωτερικό, ήταν τελούσε, βρισκόταν στο εξωτερικό και τώρα έχει γίνει επικεφαλής ε, του εκλογικού αυτού συμβουλίου. Και εγκρίνοντας το νέο εκλογικό αυτό νόμο, είδαμε ότι όλα τα πολιτικά κόμματα συμμετείχαν στη συζήτηση Υπήρξαν κάποιοι ενδιασμοί, κάποιε ανησυχίε. προσπαθήσαμε να διασκεδάσουμε αυτέ τι ανησυχίε, και πραγματικά η συζήτηση εξελίχθηκε πολύ ομαλά. Και έχουμε έπειτα και μια νομοθεσία που έχει να κάνει με τη συνεργασία για την κοινωνία των πολιτών. Και βλέπουμε ότι συμμετέχει όλο και περισσότερο η κοινωνία των πολιτών στι αποφάσει που λαμβάνονται. Και είδαμε, χάρηκα πάρα πολύ όταν είδα ότι ερχόντουσαν στο κοινοβούλιο μα πλέον πάρα πολλοί άνθρωποι, πάρα πολλοί εμπλεκόμενοι και πολλοί εκπρόσωποι τη κοινωνία των πολιτών προκειμένου να συζητήσουμε όλα αυτά τα ζητήματα που είχαν να κάνουν με τον εκλογικό νόμο. Και νομίζω ότι κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο το πολιτικό κλίμα στην χώρα μου, την Αιθιοπία. Και, όπως σας είπα, πλησιάζουν και οι εκλογές και θα ξεκινήσουν και οι πολιτικές εκστρατείες από τα διάφορα πολιτικά κόμματα και νομίζω ότι και κατά τη διάρκεια της προεκλογικής ε, εκστρατείας θα δούμε ότι τα πράγματα κινούνται πολύ θετικά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για την βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας μας και αποτελεί δέσμευση της κυβέρνησής μας, της ομοσπεδιακής κυβέρνησης, έχουμε δεσμευθεί πραγματικά προκειμένου οι επόμενες εκλογές να είναι δημοκρατικές, ελεύθερες και δίκαιες. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό αποτελεί πολύ ισχυρή δέσμευση και ελπίζω ότι η όλη προσπάθεια θα στεφθεί με επιτυχία. Δεύτερον, το ζήτημα της αρπαγής των γεών. Άμεσες ξένες επενδύσεις και αρπαγή γεών. Το ζήτημα της αρπαγής των γεών πρέπει να σας πω ότι δεν συνδέεται μόνο με τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Ακόμα και οι τοπικοί επενδυτές πολύ συχνά έχουν γεές τις οποίες δεν καλλιεργούν. Επομένως εμείς χρειάστηκε να λάβουμε κάποια συγκεκριμένα μέτρα ως προς αυτό. Δύο, είναι, δύο πράγματα είναι πολύ σημαντικά. Οι άμεσε ξένε επενδύσει είναι πολύ σημαντικέ για αναπτυσσόμενε χώρε όπω η Αιθιοπία. Αλλά ένα δεύτερο ζήτημα είναι να μπορούν πραγματικά οι τοπικέ κοινότητε να χρησιμοποιούν τι γέε. Να μπορούν να τι καλλιεργούν, να μπορούν μέσω των γεών αυτών και τη ιδιοκτησία του να δημιουργούν θέσει απασχόληση. Είναι πολύ σημαντικό να πετύχουμε την ευκταία αυτή ισορροπία. Και όπως σας είπα, ο Πρωθυπουργό ηγείται μιας επιτροπής προκειμένου να ασχοληθεί με το ζήτημα αυτό σε εθνικό επίπεδο. Το ζήτημα λοιπόν που έχει να κάνει με την ιδιοκτησία των γεωργικών εδαφών είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει ληφθεί πάρα πολύ σοβαρά υπόψη από την κυβέρνηση και νομίζω ότι θα καταφέρουμε να εξισορροπήσουμε το ζήτημα αυτό προωθώντας και τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Τώρα, ένα ακόμα ζήτημα το οποίο ετέθη. Είναι αυτό που έχει να κάνει με τις επενδύσεις που έρχονται από την Ευρώπη. Εκτιμούμε ιδιαίτερα τις επενδύσεις αυτές. Η εμπορική, η εταιρική σχέση που έχουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ σημαντική. Και θεωρώ λοιπόν ότι τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την Al-Shabaab και με την ε, επέμβαση και εμπλοκή ξένων κρατών στην Αιθιοπία, πρέπει να σας πω ότι όσον αφορά την τρομοκρατία και την αντιμετώπιση της, συνεργαζόμαστε με την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για τα ζητήματα της ασφάλειας τώρα. Εκεί προσπαθούμε να προωθήσουμε τα κοινά μας συμφέροντα. Και έτσι λοιπόν οι επεμβάσεις από τις ξένες χώρες οι οποίες υποστηρίζουν τρομοκρατικές ομάδες είναι κάτι το οποίο το καταδικάζουμε αλλά το έχετε καταδικάσει και εσείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να συνεχίσουμε τη θετική μας συνεργασία απέναντι στο φαινόμενο αυτό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα έλεγα λοιπόν ότι ακόμα και σήμερα όσον αφορά τον Νότιο Σουδάν και στη συζήτηση με τον πρόεδρο Σαλμπακύρ θέτουμε πάντα το ζήτημα της ασφάλειας διότι πολλά παράνομα όπλα καταφθάνουν από τον Νότιο Σουδάν στην Αιθιοπία και αποσταθεροποιούν τη δική μου τη χώρα. Προσπαθούμε λοιπόν να συνεργαστούμε με τις όμορες μας χώρες. Προφανώς έχουμε πολύ καλούς φίλους στην Ερυθρέα, το Σουδάν, το Νότιο Σουδάν, την Κένια, το Τζιπουτί, τη Σομαλία. Την προηγούμενη εβδομάδα σε μια συνεδρίαση στην Αντίσα Μπέμπα, στην τελετή για τα εγγένεια του νέου Προεδρικού Μεγάρου είχαμε εκπροσώπου από όλε αυτές τις φιλικές χώρες και από κοινού συνεργαζόμαστε με αυτές προκειμένου να εξαλείψουμε τρομοκρατία από το τη Αφρική. Όσον αφορά τώρα την μεταρρύθμιση του δικαστικού τομέα. Ο, η πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου ήταν ε, στο παρελθόν μια ακτιβίστρια υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των γυναικών. Τώρα, όπω σα είπα, είναι επικεφαλή του Ανώτατου Συμβουλίου. Καταβάλει πάρα πολύ σημαντικέ προσπάθειε και έχουμε και μια επιτροπή ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων στο πλαίσιο του ανώτατου δικαστηρίου που προσπαθεί να μεταρρυθμίσει την νομοθεσία που έχει να κάνει με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κατά αυτόν τον τρόπο προωθούμε και τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα εργατικά δικαιώματα και έχουμε προσπαθήσει να βελτιώσουμε και τη συνεργασία που έχουμε με την Διεθνή Οργάνωση Εργασίας. Και ξέρετε ότι ακολουθούμε ε, διαφορετική διαφορετικό ημερολόγιο αν θέλετε, οπότε φέτο τουλάχιστον για εμά θα προσπαθήσουμε να ολοκληρώσουμε όλες τι μεταρρυθμίσεις που έχουν να κάνουν με το δικαστικό μας σύστημα. Αυτό θα προωθήσει σαφώς τα μέτρα τα οποία προστατεύουν το κράτος δικαίου όσον αφορά το περιβάλλον, την παροχή ύδατο και γενικότερα την αντιμετώπιση κλιματική αλλαγή, όπω είπα στην αρχική μου παρέμβαση, εμείς θεωρούμε ότι οι πολίτες του Σουδάν και οι πολίτες της Αιγύπτου είναι πραγματικά αδέλφια μας. Συνεπώς, κατανοούμε τα προβλήματά τους και συμπάσχουμε με αυτούς. Από τεχνικής πλευράς, ο Υπουργός, ο υπεύθυνο για την παροχή ύδατος και οι ομόλογοι του από το Σουδάν, τη Σομαλία και το Τζιμπουτί συζητούν τα ζητήματα αυτά οι συζητήσει αυτέ είναι πολύ σημαντικέ και θα πρέπει να λύσουμε όλα τα τεχνικά προβλήματα. Ξέρετε ότι μερικέ φορέ ε, τα πολιτικά ζητήματα και οι πολιτικές συζητήσεις επηρεάζουν τι καθαρά τεχνικέ συζητήσει. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να επιλύσουμε τα τεχνικά προβλήματα πρώτα, έτσι ώστε να μην ζημιωθούν ούτε οι πολίτες του Σουδάνου, ούτε οι πολίτες της Αιγύπτου, είναι τα αδέλφια μας όπως σας είπα και θεωρούμε ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αυτό με ιδιαίτερη προσοχή και αποκοινούμε τις χώρες αυτές, προκειμένου να πετύχουμε μια λύση η οποία θα είναι υποφελή για όλου. Να έχουμε την καλύτερη δηλαδή διαχείριση ύδατο όχι μόνο στην Αιθιοπία αλλά και στο Σουδάν και στην Αίγυπτο. Θα επιληφθούμε λοιπόν των ζητημάτων αυτών και ελπίζω ότι σύντομα θα το λύσουμε μέσω των τεχνικών, όπω σα είπα, συζητήσεων, αλλά και μέσω τη εμπλοκή των αρμοδίων ηγετών από κάθε πλευρά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και πιστεύουμε ότι οι πολίτες της Αιθιοπίας, της Αιγύπτου, και οι πολίτες του Σουδάν είναι τα αδέλφια μας και ότι από κοινού θα πρέπει να συνεργαστούμε. Το τελευταίο ζήτημα που θίξατε έχει να κάνει με την ασφάλεια και αναφερθήκατε κυρίως στους μετανάστες από το Σουδάν, το Νότιο Σουδάν και την Ερυθρέα. Όπως το είπατε έχουμε περίπου όντω ένα εκατομμύριο πρόσφυγες από τις όμορες χώρες μας στην Αιθιοπία. Και όπως ξέρετε έχουμε και μία νομοθεσία για τους πρόσφυγες η οποία εγκρίθηκε πέρυσι από το Κοινοβούλιο μας. Σύμφωνα με τη νέα αυτή νομοθεσία, προβλέπεται ότι οι πρόσφυγες μπορούν πλέον να εργαστούν στη χώρα μας, μπορούν να έχουν άδεια οδήγηση, μπορούν να ξεκινήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα, μπορούν να ξεκινήσουν μια αγροτική δραστηριότητα. Υπάρχουν λοιπόν πλέον συγκεκριμένε επαγγελματικέ ευκαιρίε για του πρόσφυγε. Και όσον αφορά το ζήτημα τη ασφάλεια, νομίζω ότι αυτό δεν έχει να κάνει με του πρόσφυγε μόνο που έρχονται από τι γειτονικέ μα χώρε. Είναι ένα πολυδιάστατο ζήτημα. Όσον αφορά πάντω τους πρόσφυγε. θεωρώ ότι διαχειριζόμαστε καλά την κατάσταση και βέβαια είναι πολύ σημαντική και η διεθνής συνεργασία όσον αφορά τη διαχείριση του, προσφυγικού ζητήματος. Έχω στο πλάι μου και τον πρέσβη μας, ο οποίος θα ήθελε να θίξει και αυτό με τη σειρά του κάποια ζητήματα. Του δίνω λοιπόν το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Συμπρόεδρε. Σας ευχαριστώ που μας υποδεχτήκατε σήμερα εδώ. Θέλω να ε, σταθώ σε ορισμένα από τα ζητήματα που έθεσαν κάποιοι ευρωβουλευτές. Να ξεκινήσω με το, με το ζήτημα του φράγματος. Uh, για να ξεκαθαρίσω κάποιες εντυπώσεις που δημιουργήθηκαν. Δεν υπάρχει διεθνής ε, νόμος ή διεθνής συμφωνία για τη χρήση ε, των ε, υδάτων του Νείλου, στα οποία να έχει συμμετάσχει η Αιθιοπία. η Αιγύπτιοι ε, το αποκαλούν διεθνή συμφωνία, όμως είναι μια διμερή συμφωνία μεταξύ του Σουδάν και της Αιγύπτου και υπεγράφει το 1929 και το 1959. Αυτό που προσπαθούμε εμείς να κάνουμε είναι να έρθουμε σε συνεννόηση με τις 11 χώρες και το κάνουμε αυτό εδώ και 11-12 χρόνια και προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε ότι καθένα θα έχει ένα δίκαιο μερίδιο των υδάτων του Νείλου. Κατανοούμε ότι το 90% των ε, αναγκών ε, σε νερό της Αιγύπτου καλύπτονται από τον Νείλο. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να δούμε πώς τα ύδατα αυτά αξιοποιούνται και χρησιμοποιούνται εντός της Αιγύπτου. Γιατί υπάρχει τεράστια σπατάλη, υπάρχει τεράστια ποσότητα που εξαερίζεται και σχεδιάζεται και η εκτροπή των υδάτων του Νείλου σε άλλα project που αυτή τη στιγμή σχεδιάζονται ή κατασκευάζονται ήδη στην Αίγυπτο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η Αίγυπτος εξαρτάται από τον Νείλο, αλλά διαβεβαιώνουμε ότι το φράγμα της ε, Αιθιοπίας θα ε, δεν θα προκαλέσει ε, σημαντικές ε, επιπτώσεις στην Αίγυπτο. Επίσης δεν υπάρχουν προβλήματα με το Σουδάν. Οι Σουδανέζοι έχουν καταλάβει ότι θα ωφεληθούν από το φράγμα αυτό και γι' αυτό και υπήρξε μεταστροφή στο Σουδάν όσον αφορά το φράγμα. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή το Κάιρο δεν σχετίζεται μόνο με το φράγμα που κατασκευάζει η Αιθιοπία φαίνεται ότι έχουν χάσει την υποστήριξη του Σουδάν, την οποία είχαν για δεκαετίες όσον αφορά τη χρήση και την εκμετάλλευση των υδάτων του Νείλου. Εμείς λοιπόν θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις με τους ε, Αιγυπτίους, ε, ο Πρωθυπουργός Άμπε και ο Πρόεδρος Σίση κατά πάσα πιθανότητα θα συναντηθούν στην, ε, στην επόμενη εβδομάδα. το ραντεβού αυτό προσδιορίστηκε όταν ο κύριος Σίση ε, έλαβε, πήρε τηλέφωνο τον ε, Αιθίωπα Πρωθυπουργό για να τον συγχαρεί για τον Νόμπελ και νομίζω ότι ήταν πολύ θετικό το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργό μου επίσης ε, έχει ενημερώσει τον κύριο Σίση σχετικά με τις συζητήσεις που είχε η Αιθιοπία με το Σουδάν γύρω από το ζήτημα του φράγματος για την ε, τρομοκρατία στο κέρας Αφρικής και την Al-Shabaab. Η Al-Shabaab εξακολουθεί να είναι παρούσα βεβαίως. Ωστόσο η επιρροή της έχει μειωθεί. Αυτό όμως δεν θα πρέπει να μας οδηγήσει σε εφησυχασμό. Δραστηριοποιούνται ακόμη σε αρκετές περιοχές ε, της Σομαλίας Λαμβάνονται λοιπόν αντιτρομοκρατικά μέτρα κατά της Al-Shabaab και υποστηρίζεται από την Αιθιοπία η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας προκειμένου να μπορεί να σταθεί στα πόδια της. Αυτό είναι ο αγώνας και νομίζω ότι ε, είναι μια ευκαιρία σήμερα να εκφράσουμε για άλλη μια φορά την υποστήριξή μας προς την κυβέρνηση της Σομαλίας για να επιτύχει το στόχο της σταθεροποίησης και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και σε αυτό το, για αυτό το στόχο ε, χρησιμοποιούμε και αξιοποιούμε σε διαβουλεύσεις και θεωρούμε ότι η διεθνή κοινότητα επίσης πρέπει να υποστηρίξει την κυβέρνηση της ε, ε, την κυβέρνηση της Σομαλίας, όπως κάνει άλλωστε και η Αφρικανική Ένωση. Ευρωπαϊκές επενδύσεις υπάρχουν, υπάρχουν, αλλά δεν θεωρούμε ότι οι Ευρωπαίοι είναι πάτρονες της Αιθιοπίας. Ποτέ δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Γίνονται διαβουλεύσεις, διμερός με χώρες Ευρωπαϊκή Ένωση ή συνολικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου η Αιθιοπία παρουσιάζει τα έργα που θέλει να κατασκευάσει, τα ιεραρχεί όσον αφορά την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και στη συνέχεια η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει τα κονδύλια αυτά όχι μόνο για το οδικό δίκτυο αλλά και για τη δημιουργία θέσεων απασχόληση εντό τη Αιθιοπία. γιατί αυτό που βλέπουμε τα τελευταία 3-4 χρόνια και που είναι και η κατάσταση που οδήγησε στην πολιτική αλλαγή στην ε, στην ε, Αιθιοπία ήταν η ανεργία. Αρπαγή γης. Αυτό ήταν πραγματικά σημαντικό το πρόβλημα, όχι μόνο για τους ξένους επενδυτές, αλλά όπως είπε και ο Πρόεδρος, αφορούσε και αιθίωπες επενδυτές. Το πρόβλημα είναι ότι υπήρξαν πολιτικοί ε, οι οποίοι έβαζαν την υπογραφή τους σε τέτοιες αποφάσεις αρπαγής γης τα κυβερνητικά κόμματα ήταν εκείνα που ε, έδιναν ε, εκτάσεις σε ξένους και σε αιθίωπες επενδυτές. Το πρόβλημα είναι ότι πρώτον οι αποφάσεις δεν λαμβάνονταν ολοκληρωμένα, δεν εφαρμόζονταν ε, ολοκληρωμένα και δεύτερον οι επενδύσεις αυτές δεν δημιουργούσαν θέσεις απασχόλησης γιατί αν δεν δημιουργούνται θέσεις απασχόλησης τότε ε, δεν θα αυξηθεί και το ΑΕΠ και χωρίς αύξηση του ΑΕΠ, χωρίς αύξηση της απασχόλησης δεν μπορεί προφανώς να υπάρξει ε, μέλλον κοινωνικά, πολιτικά για την ε, χώρα μας. Ευχαριστώ πολύ. Uh, uh, Πρόεδρος Τομπέ, ευχαριστώ. Θέλω να πω δύο λόγια για να προσπαθήσω να κλείσω αυτήν την ε, συζήτηση. Θα ήθελα ιδιαίτερα να αναφέρω ότι πιστεύω πως οι απαντήσεις σας, κύριε ε, Πρόεδρε του Κοινοβουλίου, είναι ε, ακριβώς δείχνουν ότι μπορεί πορεία προς τις ελεύθερες δημοκρατικές εκλογές αλλά και την προσήλωσή σας σε αυτά. Ε, σε αυτή την πορεία. Ε, βεβαίως, ε, οι ερωτήσεις των πολιτικών ομάδων ήταν πολύ καλές και τις απαντήσατε ευθέως. Μιλήσαμε για, ζεστά, για καυτά θέματα όπως αρπαγή γης, δημιουργία θέσεων απασχόλησης, την κατάσταση με τους ΣΕΜΠΑΒ και την τρομοκρατία την κλιματική αλλαγή και βέβαια τη συσχέτιση όλων αυτών με την αναπτυξιακή πολιτική και την ασφάλεια. Πιστεύω πως ε, υπάρχει μια θετική, πως μάλλον βρισκόμαστε σε μια θετική πορεία αυτή τη στιγμή. Σημαντική για την Αιθιοπία αλλά και για ολόκληρη την ε, Αφρική. Αυτό το θετικό, η θετική όθεση λοιπόν είναι κάτι το που εμείς βλέπουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ήθελα να πω και εσείς είπατε πως πρόκειται για μία συνεργασία, συνεργασία που ακριβώς έτσι το βλέπουμε και εμείς από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ας προσπαθήσουμε να ε, κοδομήσουμε πάνω σε αυτή τα, τα επιτεύγματα. Θα σας δούμε στην Αντίσα Πέμπα. Σας ευχαριστώ πολύ για τη σημερινή ανταλλαγή απόψεων.